την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και των Φιλελευθέρων. Έχω λάβει τις εξής αιτήσει. Ο δυστυχώς οφείλω να σας τις αναγνώσω, διότι μέχρι αύριο δεν θα διαθέτετε πρακτικά και τα επόμενα πρακτικά θα τα βρείτε στο Στρασβούργο. Επομένως, μπορώ μόνο να σας τα αναγνώσω. Έτσι με έχουν ενημερώσει για να είναι ισχυρή, ισχυρός ο διορισμός. Βεβαίως θα τα βρείτε αυτά στο πρακτικό της συνεδριάσεως. Επειδή όμως δεν θα υπάρχει ακόμη αυτό αύριο, σας εξηγώ περί τίνος πρόκειται. Η Καρολίνα Πουνσέλ πηγαίνει στη βιομηχανία, δηλαδή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή ε, Βιομηχανίας, καθώς και στην Ισομερή Συνέλευση ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δε κύριος Νίλσον αντικαθιστά